you, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων ζήτησε να λάβει περαιτέρω πληροφορίες από τον υποψήφιο Επίτροπο κύριο Χιλ ώστε να περατωθεί η αξιολόγησή της υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίτροπος έχει δώσει απαντήσεις σε μια σειρά πρόσθετων γραπτών ερωτήσεων. Και στη σημερινή συνεδρίαση θα έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων, μια πρόσθετη ακρόαση για τα θέματα αυτά που ήταν το αντικείμενο των ερωτήσεων ώστε να υπάρξουν διευκρινήσεις που δόθηκαν γραπτά. Έχουμε μονάχα μια μισή ώρα για την ακρόαση αυτή, την πρόσθετη ακρόαση. Θα ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν την αρχή των ε, χρονοθυρίδων τριών λεπτών και υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι ο στόχος σημερινής ακρόασης είναι να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα τα οποία ηγέρθησαν στις πρόσθετες ερωτήσεις μας. Είναι λοιπόν για τις πρόσθετες αιτήσει διευκρίνησης, όχι για γενικά θέματα. Δίνω λοιπόν <clears throat> καταρχήν το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο κύριο Χιλ για την εισαγωγική του παρέμβαση 10 λεπτών και μετά θα έχουμε 24 ε, ερωτήματα, 3 λεπτών το καθένα, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο για την απάντηση. Και στη συνέχεια ο υποψήφιος επίτροπος έχει 3 λεπτά για μια καταληκτική παρέμβαση. <clears throat> Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και στο διαδίκτυο και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χιλ για την ε,